Όπως γνωρίζετε, την Τετάρτη πρωί μετά από την παρουσίαση του προγράμματος της Βουλγαρικής Προεδρίας Εξονόματος του Πρωθυπουργού της χώρας Μπόρισοφ θα γίνει η πρώτη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, στη διάρκεια της οποίας θα μιλήσει ο Τίσακ ε, που είναι μια, ένα πολύ σημαντικό ραντεβού για μας και θα είναι μια, η πρώτη από μια ολόκληρη σειρά πολυάριθμων ε, επαφών με τους ε, Πρωθυπουργού που θα τοποθετήσουν το Ευρωκοινοβούλιο στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της Ένωσης. Για να έχουμε πιο αυθόρμητη και διαδραστική συζήτηση, αποφασίσαμε για αυτή τη συζήτηση να ξεκινήσουμε ένα νέο φόρματ που προβλέπει αυθεντικό catch the eye, ώστε κάθε ευρωβουλευτή που το επιθυμεί να μπορεί να ζήσει το λόγο και να έχει την δυνατότητα να εκφραστεί. Βεβαίω, για θέματα χρόνου δεν θα μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι ε, όσο γίνεται πιο δίκαιο και να σεβαστώ την ε, ποικιλομορφία που υπάρχει στην ε, Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, παραμένει γεγονό ότι το ΚΑΣΔΕΗ θα, θα ανταποκρίνεται και στο βάρο και τον αριθμό κάθε ομάδα. Και ευχαριστώ τον Τίσακ που δέχτηκε να συμμετέχει σε αυτό το καινοτόμο, την καινοτόμα διαδικασία συζήτηση. Άρχεται λοιπόν επισήμω ε, η Σύνοδος και τα πρακτικά της περασμένης Συνόδου έχουν διανεμηθεί. Ε, ε, υπάρχουν παρατηρήσεις. Τα πρακτικά εγκρίνονται. Μετά από την παρέτηση του κυρίου Γιώσου Βαρίστια Μπαούνσε, το κοινοβούλιο